ότι χρειάζεται για να καταπολεμηθεί, καταπολεμηθούν αυτά τα αρνητικά έτσι, συναισθήματα. Επίσης, είμαι ευγνώμων για την πρωτοβουλία για την Αφρική. Έτσι όπως λέμε σε ωραία γερμανικά υπήρξε μια, ένα high level group, μια συνάντηση υψηλού επίπεδου στην Βιέννη με τους Αφρικανούς ομολόγους μας ε, γιατί θα πρέπει να υπάρξει μια διασφάλιση του αφρικανικού μέλλοντος. Αλλιώς δεν θα υπάρξει διασφάλιση του ευρωπαϊκού μέλλοντος. Αυτό ήταν λοιπόν το σημαντικό μήνυμα της Αυστριακής Προεδρίας ε, προς την Αφρική. Και ήταν πολύ σημαντικό. Συνολικά λοιπόν, με την εξαίρεση που ανέφερα, είχαμε μια επιτυχημένη Προεδρία και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Καγκελάριο, την κυβέρνηση, τον πρέσβη για τα όσα έκαναν και τις επιτυχίες που στην αρχή της Προεδρίας δεν νομίζαμε ότι θα συμβούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν. Να περάσουμε στου εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Ε, παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο αγόρευσης, γιατί όπως ε, ξέρετε έχουμε και την παρενική συνεδρίαση για την 20η επέτειο του ευρώ. Τώρα ο κύριος Βέμπερ, που είναι πρόεδρος ε, του ΕΛΚ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γιούνκερ, κύριε Καγκελάριε, κύριε Πρέσβη, αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε στον απολογισμό της Προεδρίας του Συμβουλίου και εμείς ε, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για, την έντυπωση, για τον εντυπωσιακό αυτό απολογισμό της ε, Προεδρίας σας για τα όσα καταφέρατε αυτούς τους έξι μήνες για το μέλλον της Ευρώπης. Ε, ειλικρινά σας λέω, καμιά φορά είναι κρίμα το ότι οι δημόσιες συζητήσεις για την Ευρώπη αφορούν πάντα τις κρίσεις, πάντα τα προβλήματα που υπάρχουν και δεν καταφέρνουμε να συζητήσουμε τα θετικά τα όσα καταφέρνουμε, αυτά τα οποία ενισχύουν την Ευρώπη. Είναι κρίμα. Έτσι, ε, βεβαίω ε, ζούμε ως πολιτική, αλλά αυτό το αποδεικνύει ιδιαίτερο η Αυστρική Προεδρία. Ο πολιτικός απολογισμός ήδη έγινε. Ως ομάδα του ΕΛΚ θα θέλαμε να τονίσουμε τα θέματα της ασφάλειας, το Ταμείο Άμυνας, ε, ο τομέας των μη επανδρομένων αεροσκαφών επίσης ε, προσφέρει ε, πάρα πολλές ε, προοπτικές. Έχουμε το θέμα της ευημερία. Επιτύχαμε εκεί πέρα σημαντικές προόδους. Τον έλεγχο των επενδύσεων κατ' σημαντικό. Η συμφωνία με την Ιαπωνία επίσης έκλεισε και όσον αφορά τις χρεώσεις περιαγωγής, ε, το καταφέραμε όπως επίσης και για τα τραπεζικά εμβάσματα και την απαγόρευση των πλαστικών και το διοξίδιο του άνθρακα. Είχαμε αρκετές επιτυχίες ε, και αν μπορούσαμε να το μεταδώσουμε αυτό στον κόσμο θα πήγαινε και καλύτερα η Ευρώπη. Σημαντικό είναι επίσης το ότι ξεκίνησαν πολιτικές ε, συζητήσεις γιατί βεβαίως είναι κάποια διαχείριση η Προεδρία αλλά πρέπει να δώσει και κατευθύνσεις στο πρώτο άτυπο συμβούλιο στο Σάλτσμπουργκ κατέθεται το ζήτημα της προστασίας των εξωτερικών συνόρων. Για εμάς είναι κεντρικό ζήτημα, είναι προϋπόθεση για οποιαδήποτε άλλη συζήτηση στον τομέα της μετανάστευσης. Το θέμα της δικαιοσύνης με τον ψηφιακό φόρο. για να πληρώσουν αυτό που τους αναλογεί και οι μεγάλη όμιλη του διαδικτύου. Σας συγχαίρω λοιπόν γι' αυτό. Αυτό νομίζω ωφέλησε την Ευρώπη και η συζήτηση βεβαίως θα ανέφερε ο Ζαν για το εάν είμαστε στην Ευρώπη σε μια ήπειρο που μιλάμε ξανά σοβαρά για βία κατά των Εβραίων πρέπει αυτό να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα το θέμα δηλαδή του αντισημιτισμού και αυτά τα οποία μας είπαν οι εβραϊκές ενώσεις πρέπει να μας ανησυχήσουν. Και το βασικό μήνυμα εδώ πέρα είναι ποτέ ξανά. Σας συγχαίρω λοιπόν. Τέλος θα ήθελα να πω πως η Αυστρία είναι οπωσδήποτε ε, ισχυρή χώρα με μια ισχυρή κυβέρνηση και οι πολίτες ε, νομίζω το είδαν όπως και εγώ ότι ήταν υπερήφανοι που είχαν για ένα εξάμεινο την Προεδρία της Ευρώπης ε, και ήταν ε, πάρα πολύ θετικό και αυτό το οποίο παραμένει είναι η επικοδομητική συνεργασία, η ηγεσία που επιδείξατε και η συνένεση που ε, οδηγούν όλα αυτά σε πρόοδο στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν. Επόμενη ομιλήτρια, κυρία Ροντρίγκε από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Καγκελάρη, η Αυστριακή Προεδρία ξεκίνησε με ένα σημαντικό μότο, μια Ευρώπη που προστατεύει. Και πράγματι χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που να προστατεύει. Όμως θεωρούμε την, ότι η Αυστριακή Προεδρία παρουσίασε περισσότερα αποτελέσματα, μια άλλη Ευρώπη, μια Ευρώπη φόβων ε, και μια Ευρώπη υπεναχωρήσεις και εγωισμών ε, και το λυπούμαστε γι' αυτό γιατί χρειαζόμαστε μια Ευρώπη με μεγάλες ε, φιλοδοξίες έτσι ώστε να μπορούμε να δώσουμε και την απαραίτητη αλληλεγγύη. Αυτό ξεκίνησε με τη δραματική κατάσταση για τους πρόσφυγες. Θα μπορούσαμε να είχαμε ταχείες επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής ασύλου. Όμως ε, είδαμε διάφορα τραγικά γεγονότα στη Μεσόγειο και λυπούμαστε γι' αυτό. Η Ευρώπη θα πρέπει να καθορίσει μια πλήρη πολιτική για το μεταναστευτικό για να μπορεί να διαχειριστεί τη μετανάστευση, μια έφτακτη μετανάστευση, γιατί χρειαζόμαστε τη μετανάστευση. Αντιθέτως όμως μπλοκάρουμε κάποια κύρια τμήματα αυτής της μεταναστευτικής πολιτικής και κατόπιν λυπούμαστε για το τι συνέβη με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση γιατί επικυρώθηκε από τις περισσότερες χώρες του κόσμου και είδαμε ότι στο Μαρακές κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην κυρώνουν το σύμφωνο αυτό από την ηγεσία της αυστριακής κυβέρνησης. Και πάλι εκφράζουμε τη λύπη μας γι' αυτό και δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Όμως αυτή η έλλειψη φιλοδοξίας και αλληλεγγύης έχει συνδεθεί και με τους πολίτες. Γιατί για να δούμε τι γίνεται με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα, τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία που έχουμε. Η Αυστριακή Προεδρία θα μπορούσε να έχει παρουσιάσει ταχύτερα αποτελέσματα για όλο το σύνολο των οδηγιών που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του κοινωνικού πυλώνα και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς ήταν δυνατό η Αυστριακή Προεδρία να αναβάλει μια συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών. Βιαζόμαστε, κύριε Καγκελαρή, για να εφαρμόσουμε αυτόν τον πυλώνα και να τον καταστήσουμε πραγματικότητα. Και κατόπιν έχουμε τις σημαντικές διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ναι, είναι κάτι απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις στην Ευρώπη, και για να έχουμε και ισχυρή δέσμευση Ω προ τη συνοχή, απογοητευτήκαμε που στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίστηκε ότι η τελική συμφωνία θα πρέπει να ληφθεί, να γίνει τον φθινό, το φθινόπωρο. Έχουμε τις προϋποθέσεις να καταλήξουμε σε μια βασική συμφωνία νωρίτερα. Και δεν κατανοούμε γιατί η Αυστριακή Προεδρία δεν ήταν ικανή να παρουσιάσει ένα πιο φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις αυτές. Κατόπιν, είχαμε μια άλλη ευκαιρία για τη μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης. Πρόκειται για κάτι που περιμένουμε εδώ και χρόνια. Οι λύσει είναι επιτάπητος. Μπορεί να είμαστε κοντά σε μια συμφωνία που θα μας βοηθήσει να ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση και να δημιουργήσουμε ένα προπολογισμό για την Ευρωζώνη. Κάτι που έχουν όλε οι νομισματικέ ενώσει ε, παγκοσμίω. Έχουν προπολογισμό. Όμω και πάλι η Αυστρική Προεδρία δίσταζε. Και αυτό είναι ένα ε, ζωτικό στοιχείο για να έχουμε εκ νέου συνοχή στην Ευρωζώνη και να καταπολεμήσουμε τις αποκλίσεις ε, σε αυτό το σημαντικό τομέα του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος και κατόπιν φορολογική δικαιοσύνη. Ναι, χρειαζόμαστε ένα νέο ψηφιακό φόρο για τις ψηφιακές υπηρεσίες και θα πρέπει ταχύτερα να τον υλοποιήσουμε. Έτσι, λοιπόν, από τη δική μας σκοπιά, κύριε Καγκελάρε, η Αυστριακή Προεδρία έχασε κάποιες σημαντικές ευκαιρίες για να οικοδομήσει μια πιο ισχυρή Ευρώπη που χρειαζόμαστε αυτή τη σε αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία. Γιατί βλέπουμε μια νέα κίνηση ιδεών και ε, βλέπουμε εδώ ότι ε, βλέπουμε εγωισμούς, ε, ακροδεξιά κινήματα και εγκλωβισμούς και απέναντι σε αυτό έχουμε την εξής επιλογή, είτε θα συμμαχίσουμε μαζί τους και θα κάνουμε κάποιες εκχωρήσεις τα κινήματα αυτά ή θα παρουσιάσουμε μια πλήρη εναλλακτική, μια ισχυρή φιλόδοξη Ευρώπη που να μπορεί να παρέχει αλληλεγγύη. Έτσι λοιπόν αυτή είναι η οδός που πρέπει να ακολουθήσουμε εμείς, θεωρούμε, οι σοσιαλιστές και δημοκράτες και θα πρέπει να κινηθούμε σε ένα νέο στάδιο που ε, τέτοιες ηγεσίε θα αναδυθούν στην Ευρώπη. Αυτό είναι το δικό μας μότο, κύριε Πρόεδρε. Επόμενο για του συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ, ο κύριο Ζάχραντιλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λυπή Πρόεδρε, κύριε Καγκελάρη. Γενικώ η Αυστριακή Προεδρία διοργανώθηκε σωστά, ήταν αποτελεσματική και καλά συντονισμένη. Και αυτό γιατί η Αυστρία είναι μια χώρα η οποία λειτουργεί εύρυθμα. Ε, καλύψατε πολλά θέματα στην ομιλία σας. Εγώ θα επιλέξω μόνο μερικά μεμονωμένα σημεία, ξεκινώντας με τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Πρέπει να σας πω ότι πραγματικά ήταν ε, σχεδόν διασκεδαστικό να ακούσουμε μια διαφορετική σκοπιά από την πλευρά της Προεδρίας και της Καγκελαρίας από ότι στο παρελθόν συνέβαινε. Είπατε ξεκάθαρα κάτι που άλλοι πολιτικοί δίσταζαν να πούν καθαρά, ότι η Ευρώπη δεν είναι ούτε έτοιμη ούτε πρόθυμη να δεχτεί ε, αλλεπάλληλα κύματα μεταναστών. Αυτό θα είχε επιπτώσεις και στην ασφαλειά μας, αλλά και στην εσωτερική μας συνοχή, στις κοινωνίες μας. Και επίσης υποβάλλατε ε, προτάσεις και λύσεις, όπως την αναθεωρήση του κώδικα των συνόρων για το Σέγγεν και την ε, αρρωγή για την υποδοχή της μετανάστευσης και την αντιμετώπιση της λάθρομετανάστευσης. Σίγουρα τα μηνύματά σας αυτά ακούστηκαν από πολλούς με προσοχή, ε, ξεκάθαρα, και στην Κεντρική Ευρώπη και σε άλλες χώρες και πάλι από δείχθηκε ότι είναι πολύ σημαντικό να αναζητάτε συμβαστική λύση μεταξύ των κρατών μελών αντί να επιλέγουμε αυθαίρετες λύσεις. Όπως ε, το ατυχές ε, σύστημα επαναγκατάστασης που προώθησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κόστισε μάλλον προκάλεσε μια από τις μεγαλύτερες διενέξεις μεταξύ Δύσης και Ανατολικής Ευρώπης και σίγουρα ε, έφερε ένα νέο διαχωρισμό μεταξύ κρατών και νέων και παλαιών και των μελών. Σίγουρα η ευημερία και η ανταγωνιστικότητα τη ευρωπαϊκή οικονομία είναι κάτι που προάγατε με την ψηφιοποίηση και την κοινοτομία και είχατε δίκιο. Ενώ λειτουργεί καλά η κουλτούρα μας για τις νοφίες επιχειρήσεις. Ε, οι μεγάλοι στο χώρο αυτό έρχονται από άλλες περιοχές του κόσμου. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα στην Ευρώπη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να άρουμε τους εμπορικούς φραγμούς και θέλω να σας συγχαρώ γιατί πετύχατε τη γρήγορη έγκριση της εμπορικής ε, συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με την Ιαπωνία. Έτσι δημιουργήσαμε τη μεγαλύτερη εμπορική περιοχή καλύπτοντας το, ε, ένα, το 70% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Ελπίζουμε να προχωρήσουν οι συμφωνίες με την Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ. Και βεβαίως οι διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν επί τη Προεδρία σα θα συνεχιστούν. Αυτό είναι ευχάριστο γιατί και το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή φτάνουν στο τέλο τη θητεία του. Δεν θα πρέπει να αποφασίσουν εκ μέρου των 100 μελών ή ε, προδικάζοντα το τι θα κάνουν οι μελλοντικοί επιτροποί. Για τι εξωτερικέ μα σχέσει. Δεν θα επεκταθώ απλώς να δηλώσω ότι η Αυστρική Προεδρία είχε πραγματιστική προσέγγιση, δεν ήταν θύμα ιδεολογιών και επεδίωξε χειροπιαστά και από τα αποτελέσματα. Δηλαδή η κοινή λογική ε, υπερίσχυσε. Ε, η κοινή λογική είναι και κάτι που προσπαθεί να προάγει και η δική μου ομάδα σε αυτό το κοινοβούλιο. Επιτέλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο λόγος στον κύριο Τελίτσκα, εκ μέρους των φιλελευθέρων. Καγκελάριε, δεν είμαι βέβαιος εάν θα αντέξετε να ακούσετε κι άλλα συγχαρητήρια, γιατί ακούσατε ήδη πολλά σήμερα, οπότε θα σα απαλλάξω. Ήταν αποτελεσματική η προεδρία σα. Η Αυστρία έφερε αποτελέσματα, ε, ε, ήταν συνεπής με όσα είχε αρχικά ανακοινώσει, όμως κάθε έξι μήνες το θέμα δεν είναι εάν τα πήγε καλά απλώ η Προεδρία. Δεν θέλουμε να συζητήσουμε μόνο αυτό, αλλά και το πώ τα πήγε η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχέτω Προεδρία. Αυτό που πρέπει λοιπόν να ακουστεί σήμερα είναι ότι μιλάμε ακόμα για μια Ευρωπαϊκή Ένωση των 28, που μπορεί σύντομα να είναι 27 κράτη-μέλη. Η Προεδρία έχει το ρόλο τη να διαδραματίσει. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνη τη, αλλά μπορεί να κάνει πολλά για την Ευρώπη. Αυτό λοιπόν ήδη είναι ένα ε, καλό στόχου. Τώρα μιλήσατε για τον αριθμό των τριμερών διαλόγων και αυτό είναι ε, ένα δείγμα ε, αποτελεσματική προεδρία, αλλά να δούμε τι έγινε με την νομοθεσία που εφαρμόζεται. Είναι ε, η νομοθεσία που εγκρίθηκε αυτή που θα επιδιώξει του στόχου που ανακοινώσατε και εσεί, του τρει στόχου που αναφέρατε προηγουμένω. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Η συγγήτρια Αγγελικά ασχολήθηκε με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Δεν ήταν κακό το αποτέλεσμα, ήταν μάλλον καλό. Όμως, παρά τις διάφορες ε, διαφιλονικίες που είχαμε με τον πρεσβευτή της Αυστρίας, ε, που είχε πολύ έντονη παρουσία στου τελευταίους διαλόγου, παρόλα αυτά αντικατοπτρίζεται η έλλειψη αλλαγή νοοτροπία και κουλτούρα στα κράτη-μέλη. Ακόμα την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο τον την βλέπουν σαν ένα θέμα όπου παίζουμε ε, μεταξύ όσων θέλουν να προασπιστούν εταιρικά συμφέροντα και όσων όχι. Εδώ πρέπει να αποφασίσουμε αν είμαστε δυνατοί ή αδύναμοι. Είμαστε ο πιο αδύναμο κρίκο τη αλυσίδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αναφέρω το εξή. Ε, το, θέμα δεν είναι απλώ πόσου τρομερέ διαλόγου ε, οργανώσαμε, αλλά τι νομοθεσία εγκρίναμε και τι κατάφεραν να συμφωνήσουν μεταξύ του τα κάθε μέλη με συμβαστικέ λύσει για το επίπεδο φιλοδοξιών του. Για την ε, ψηφιακή προστασία των δεδομένων. Ε, ναι, υπήρξε πρόοδος, αλλά εγώ αν είχα το μυαλό θα μπορούσα να εφεύρω μια ε, εφαρμογή που να λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να την πουλήσω εγώ στο Silicon Valley. Αυτό θα ήθελα να κάνω. Δυστυχώ δεν έχω το μυαλό. Είναι πολλά λοιπόν που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το εμπορικό τη οικοσύστημα. Θα ήθελα λοιπόν να επικεντρωθώ σε δύο-τρία ζητήματα στα οποία θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει καλύτερα. Οπωσδήποτε και είναι και ένας γνώμονας για την Προεδρία. Το ένα είναι η ε, εσωτερική ασφάλεια. Ναι, είχατε καλά εξισορροπημένη προσέγγιση, όμως να το παραδεχτούμε. Ακόμη έχουμε μπλοκάρισμα στο Συμβούλιο για πολλέ προτάσει, οι οποίε εκκρεμούν. Είναι σε τέλμα. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την τωρινή κρίση και τα τωρινά προβλήματα ε, με αυτέ τι λύσει. Θα έχουμε σοβαρά προβλήματα αν αυτά ενταθούν για τον προπολογισμό. Και πάλι Τεράστια πρόοδο επετεύχθη. Δεν μπορώ να πω. Όλα τα κουτάκια που έπρεπε να συμπληρώσετε πήραν τικ. Αλλά πώ συμπληρώθηκαν. Όπω είπε ο κύριο ε, Ζάχραντιλ, ε, να τα αφήσουμε αυτό στην επόμενη θητεία. Όχι, ε, εξελέγημεν, για ολόκληρη τη θητεία εμεί, για, την, για ολόκληρη την πενταετία. Άρα, όταν μιλάμε για την συνοχή, αν μιλάμε για του γεωργού και βλέπουμε ότι καθυστερούμε, αυτό επηρεάζει τι δουλειέ του, επηρεάζει το πώ θα πάνε. Οπότε ο προπολογισμό είναι ένα δείγμα για το πώ ε, μα αντιλαμβάνονται απ' έξω. Και δεν είναι κατηγορία για την Αυστρία αυτό. Είσαστε ρεαλιστέ, ναι, και εγώ είμαι κατά τη οποιασδήποτε σπατάλη και διασπάθηση ε, κονδυλίων. Όμω με τι νέε προκλήσει που έχουμε μπροστά μα δεν μπορούμε να συνεχίσουμε απλώ να θεωρούμε κάποιε πολιτικέ και ε, να μην αυξάνουμε πουθενά τον προπολογισμό. Και εν τέλει, με αυτέ τι παρατηρήσει, παρόλα αυτά να πω ότι η δουλειά σα ήταν καλή, αλλά ω Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη δεν είμαστε στο ύψο των προσδοκιών των συμπολιτών μα σε πολλά ζητήματα μένουμε πίσω. Ευχαριστώ. Τώρα, στην κυρία Σκακέλερα από τους Πρασίνους θα δώσω το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ δυστυχώς κύριε Κούρτς δεν μπορώ να συνταχθώ με τους προλαλήσαντες. Τι απέμεινε τελικά από την Αυστριακή Προεδρία δεν προχώρησαν. Πολλές νομοθετικές προτάσεις κόλλησαν στο Συμβούλιο, αλλά αυτό το οποίο πραγματικά θα μας μείνει σε εμά και εκτός από την αίθουσα στους τελευταίους έξι μήνες είναι η πραγματικά λυπηρή υπόκλησή σας στον πρόεδρο Πούτιν αλλά και το ότι αρνηθήκατε να συνυπογράψετε το σύμφωνο του ΟΗΕ για την μετανάστευση ειδικά η αυστριακή κυβέρνηση αρνήθηκε να υπογράψει αυτή την προσπάθεια τόσων πολλών κρατών του κόσμου για να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Και πραγματικά ενώ καταβάλατε κι εσείς προσπάθεια στο να συνταχθεί, να παριστάνετε μετά ότι είναι του σατανά, είναι ανεξήγητο. Ε, πολλώσατε λοιπόν και μπήκατε μόνοι σας ε, στην ε, ακροδεξιά γωνία όπως ο Τραμπ και ο Όρμπαν. Και εκεί πέρα μας βλάψατε όλους, ε, ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Είναι έτσι ξεκαθαρό ότι η κυβέρνησή σας έκανε πραγματικά ό,τι ήθελε ενώ υπήρχε διακριτική μεταχείριση πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το να περικοπούν κάποια οικογενειακά βοηθήματα. Τέλος πάντων. Στα θετικά όμως ε, δεν υπάρχουν τόσα πολλά στους τελευταίους ε, έξι μήνες ούτε στην καταπολέμηση της ε, φοροαποφυγής και του φορολογικού dumping ούτε σε ζητήματα διοξιδίου του άνθρακα. Εκεί πέρα απλά ήσασταν ε, παρακολούθημα της ε, γερμανικής ε, αυτοκίνητοβιομηχανίας. Δεν έγινε και τίποτα και στην Frontex. Ούτε καν στην Frontex αναβλήθηκαν τα πάντα και υποτίθεται ότι ήταν προτεραιότητα της Αυστριακής Προεδρίας. Όσον αφορά Όντω, τα πλαστικά μιας χρήσης κάτι έγινε και εδώ πέρα πρέπει να επενέσω τους υπαλλήλου σας και νομίζω ότι η μεγαλύτερη κατάκτηση της ε, Προεδρίας σας ε, ήταν ε, ότι κερδίσατε στο Κατοβίτσε το βραβείο που δώσαμε για το απολύθωμα της ημέρας. Αλλά η κοινωνία των πολιτών στην Αυστρία είναι διαφορετική. Πάρα πολλοί κόσμος εμπλέκεται, βγαίνει στους δρόμους κατά του ρατσισμού και κατά Τη μείωση του κοινωνικού κράτου. και ελπίζω ε, να κερδίσουν αυτοί οι άνθρωποι στην Αυστρία και στις ε, ευρωεκλογέ. γιατί η Ευρώπη χρειάζεται μια Αυστρία ανοιχτή στον κόσμο και ολόκληρη η Ευρώπη χρειάζεται μια κοινωνία των πολιτών όπως η δική σας ε, κατά του διχασμού και υπέρ της κοινωνικής συνοχής. Σας ευχαριστώ. Από την ΚΟΕ, ο κύριος Παπαδημούλης έχει το λόγο. Κύριε Κούρτς, λυπάμαι, αλλά θα σας απογοητεύσω. Δεν συμμερίζομαι το κλίμα των αυτοεπένων και των συγχαρητηρίων. Θεωρώ ντροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Αυστρία ως προεδρεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρνήθηκε να υπογράψει το σύμφωνο του ΟΗΕ για τη μετανάστευση στο Μαρακές. Ένα σύμφωνο που υπέγραψαν 150 χώρες από όλο τον πλανήτη μετριοπαθές, ισορροπημένο, στην προετοιμασία του οποίου είχατε συμβάλει. Και θέλω να μας απαντήσετε στη δευτερολογία σας. Γιατί ντροπιάσατε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προεδρεύων αρνούμενος να βάλετε την υπογραφή σας σε αυτό το κείμενο. Δεν σας τα λέω μόνο εγώ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Σας τα είπε πιο ευγενικά, πιο κομψά και ο κύριος Γιούνκερ που ανήκει στην πολιτική σας ομάδα. Και επίση, δεν κάνατε τίποτα για τον ευρωπαϊκό κοινωνικό πυλώνα. Δεν κάνατε τίποτα ουσιαστικό για να προωθήσετε το πακέτο μεταρρύθμισης του Δουβλίνου, στο οποίο έχουμε συμφωνήσει εδώ και καιρό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν. Το καθυστερείτε και το μπλοκάρετε. Για την πανευρωπαϊκή εγγύηση καταθέσεων, το περίφημο EDIS, και πάλι αναβλητικότητα και καθυστέρηση με αποτέλεσμα να μην ολοκληρώνεται η τραπεζική ενοποίηση. Για την φορολόγηση των γιγάντων του διαδικτύου. Τίποτα συγκεκριμένο. Για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η δουλειά σας ήταν να επιταχύνετε τις συγκλήσεις για να έχουμε μια συμφωνία πριν από τις ευρωεκλογές, γιατί η αναβολή λήψης αποφάσεων σε αυτό το θέμα κάνει ζημιά στην ευρωπαϊκή οικονομία. Πολύ φοβούμε ότι η συγκυβέρνησή σας με ένα κόμμα της άκρας δεξιάς, το οποίο ιδρύθηκε από οπαδούς των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σας επηρεάζει καθοριστικά. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ανησυχητικό το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά τις ευρωεκλογέ μια τέτοια συμμαχία δεξιάς άκρας δεξιάς. Επειδή σας επέκρινα πολύ, θα κλείσω με μια θετική αναφορά. Θεωρώ θετικό ότι και εσείς και ομόφωνα το Συμβούλιο και ομόφωνα η Κομισιόν και όλες οι πτέρυγες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στηρίζουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι μια συμφωνία θετική για την Ελλάδα, θετική για τη βόρεια μακεδονία θετική για τα βαλκάνια θετική για όλη την ευρώπη είναι μία από τις καλές ειδήσει που έχουμε δυστυχώς λίγες αυτή την περίοδο και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι τις επόμενες ημέρες η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση Τσίπρα, είναι αποφασισμένη να κυρώσει τη Συμφωνία των Πρεσπών στο Κοινοβούλιο της Αθήνας παρά την αντίδραση την μικροπολιτική την δημαγωγική των κομμάτων της νέας δημοκρατίας και του πασόκ που σε αντίθεση με τις πολιτικές ομάδες του ελκ και των σοσιαλιστών αντιπολιτεύονται και αρνούνται την κύρωση της συμφωνίας των πρεσπών. Σας ευχαριστώ για την Ευρώπη των Ελευθεριών και της Άμεσης Δημοκρατίας, ο κύριος Μόιτεν. Πρόεδρε, κύριε Γιούνκερ, κύριε Κούλτς. Πρώτα απ' όλα να σημειώσω τρία θετικά πράγματα στα πρακτικά. Πρώτα απ' όλα, η γη συνεχίζει να γυρίζει. Δεύτερον, δεν έγιναν πόλεμοι. Και τρίτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να γραφειοκρατικοποιείται. Και όλα αυτά παρά την πρεμιέρα αυτή που είχαμε. Οι λεγόμενοι δεξιοί λαϊκιστές συμμετείχαν για πρώτη φορά σε μια κυβέρνηση και αυτή είχε την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτό δείχνει πω κάποια πράγματα αλλάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα δραστικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα είναι μια διαφορετική Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι ήταν πριν από την Αυστριακή Προεδρία. Γιατί υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο συνέβη για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά η Προεδρία του Συμβουλίου δεν ε, αισθάνθηκε την ανάγκη να είναι η πιο συγκεντρωτική ε, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν ρεαλιστική χωρίς να προωθεί τον συγκεντρωτισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το σύμφωνο του ΟΗΕ για τη μετανάστευση. Εμείς το θέσαμε αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη και τολμώ να ισχυριστώ ότι δεν θα είχε κυριαρχήσει στη συζήτηση στην Ευρώπη εάν δεν υπήρχε η Αυστριακή κυβέρνηση η οποία ήταν πραγματικά αποφασισμένη και στις δηλώσεις της. Η Αυστρία πραγματικά κατάφερε να ξεχωρίσει από τους yes και έτσι κατάφερε να υπάρξει μια δημόσια συζήτηση για αυτό το καταστροφικό σύμφωνο. Σας ευχαριστώ λοιπόν κύριε Κούρτς. Γι' αυτό θεωρώ ότι η Αυστριακή Προεδρία μία μέρα θα θεωρηθεί ένα σημείο καμπής στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είμαι ο μόνος, νομίζω, ο οποίος Αντιλαμβάνεται την δύναμη που έχει μία προεδρία του Συμβουλίου. είμαι σίγουρος ότι σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλες προεδρίες του Συμβουλίου, το αυστριακό παράδειγμα. Κυρίες και κύριοι, μία μικρή αντίσταση κατά της ε, ακόμα κυρίαρχης τάσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σας καθιστά αντιευρωπαίους. Αντιθέτως, το να μην είστε γέσμεν και να λέτε συνεχώς αμήν και οσανά είναι υποχρέωση των κρατών μελών. Χρειαζόμαστε επιτέλους κάποιες δικλείδες ασφαλείας που θα λειτουργούν, να ακουστεί και κάποιο όχι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπό την ηγεσία Κομισιών και Κοινοβουλίου λειτουργεί ως υπερκράτος. Αυτό το όχι θα το ακούμε συχνότερα στο μέλλον και θα κάνει καλό στην Ευρώπη. Αυτό προβλέπω εγώ. Ευχαριστώ. Στην Ευρώπη των Εθνών και ε, των Ελευθεριών, ο ε, συνάδελφε Λίνσκι έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Σαν Αυστριακός θα ήθελα να ξεκινήσω ευχόμενος στον καγκελάριό μα τον κύριο Σεμπάστιαν Κόλτ. καθώς ήρθε, το καλώ ήρθε στο Κοινοβούλιο και στον κύριο Κουρτ και θα ήθελα να διαβιβάσει ευχαριστή στην αντιπροσωπεία μου ε, και να διαβιβαστούν αυτέ οι ευχαριστήσεις και προ την κυβέρνηση. Αυτή η Προεδρία του Συμβουλίου, η Αυστριακή, ήταν πολύ επαγγελματική, πάρα πολύ επαγγελματική και υποδειγματική για όλους εκείνους που προσπαθούν να κατηγορήσουν ή να αναμαυρώσουν την Αυστριακή Προεδρία πρέπει να πω ότι πρέπει να πούμε στους σοσιαλδημοκράτες ότι έχουμε και του, έχετε τους Ρουμάνους σοσιαλδημοκράτες στην ομάδα σας και πρέπει να το θυμηθείτε αυτό. Και αν βλέπετε τα θέματα διαφθοράς και άλλα συναφή θέματα, να θυμηθείτε ότι δεν είσαστε ε, ε, και πολύ δεν είσαστε τόσο αθώοι ώστε να κατηγορείτε άλλους. και οι πράσινοι συνεχώς διαμαρτύρονται για το κόμμα ελευθεριών, ε, της ελευθερίας στην Αυστρία. Αλλά εκείνο αποφάσισε, αυτό το κόμμα αποφάσισε στην Αυστρία να εργαστεί σκληρά για το θέμα των αποζημιώσεων και τη συνεργασία με το Ισραήλ. Πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε αντικειμενικοί και να μην ε, απαγγέλουμε κατηγορίες κατά άλλων κομμάτων. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι δεν μπορούσε να κατανοήσει γιατί η Αυστρία δεν επικύρωσε ε, το σύμφωνο του ΟΗΕ για τη μετανάστευση. Διότι υπήρχε μια τέτοια δημοκρατική πλειοψηφία εντός της κυβερνήσεως και του Κοινοβουλίου που ήθελε να συνεχίσουμε να καθορίζουμε εμείς τη μεταναστευτική μας πολιτική, εμείς οι ίδιοι και δεν θέλαμε να κυρώσουμε ένα μη δεσμευτικό σύμφωνο που τελικά θα κατέληγε από μη δεσμευτικό να καταλήξει, θα γινόταν δεσμευτικό. Νομίζω ότι είναι σωστό να μην αγνοήσουμε και τη θέση του ανωτάτου δικαστηρίου μας. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Αυστρίας στο Συμβουλίο, το θέμα της επικουρικότητας ε, στηρίχθηκε δεόντω. Έγινε μια διάσκεψη στο Μπρέγκενς όπου άνοιξε το δρόμο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και έλεγε ότι πρέπει να επανέλθουμε σε εθνικές αποφάσεις και είναι καλύτερο να λαμβάνονται οι αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο. Η Προεδρία του Συμβουλίου, η Αυστριακή, υπήρξε έξοχη. Και ελπίζω ότι μια τέτοιου είδους Προεδρία θα είναι υπόδειγμα για το μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ την αστική κυβέρνηση. Λόγω έχει ο κύριο Ουγιασδόφσκι από του μια Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καγκελάριο κύριο κουρτ για την πολύ ρεαλιστική και πραγματιστική αυστριακή προεδρία που άσκησε. Γιατί είναι πολύ πιο θετική αυτή η στρατηγική γευνακή για την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη στρατηγική της περισσότερης ολοκλήρωσης και της πιο περισσότερης και πιο παρούσης Ευρώπης. Ιδιαίτερα στα θέματα της οικολογίας, της προστασίας της αγοράς απέναντι στο, στα μεγαθύρια του ίντερνετ. Ήταν πολύ σημαντικά επιτεύγματα της Αυστριακής Προεδρίας. Τα παρουσιάσατε και στην ομιλία σας. Μάλιστα υπήρξε μεγάλη διαφορά με τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής ε, στη συζήτηση για τη μεταναστευτική πολιτική. Και αυτέ οι διαφορέ μεταξύ ε, Κομισιόν και Συμβουλίου δείχνει πόσο πιο λογική ήταν η Αυστριακή Προεδρία, γιατί η αλληλέγγυα πολιτική απέναντι στου μετανάστες θα πρέπει να είναι υπεύθυνη πολιτική και ρεαλιστική πολιτική, σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που διέπραξε μείζον σφάλμα ε, επιβάλλοντας το σύστημα των ποσοστώσεων για την υποδοχή μεταναστών κάτι που μείωσε την εμπιστοσύνη του λαού προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οδήγησε σε μία αύξηση και σε έξαρση του λαϊκισμού, της δημαγωγίας. Ε, θα πρέπει να είμαστε συνετοί, σόφρονες, να ασκούμε μια αλληλέγγυα πολιτική που θα είναι όμως πρώτα απ' όλα ρεαλιστική. Και καλό θα ήταν να αναλογιστούμε την πολύ θετική εμπειρία της Αυστριακής Προεδρίας από την άποψη αυτή. Επίσης, συμφωνώ να καταπολεμήσουμε τον αντισημιτισμό, όπως είπε ο καγκελάριος Κούρτς, και πιστεύω ότι θα ε, τεθούν σωστά θεμέλια, ώστε να γίνει μια ευαισθητοποίηση υπέρ της ανεξιθρησκείας και της ελευθερίας της ε, θρησκευτικής ε, πεποίθησης. Και κυρίως να προστατεύσουμε τους χριστιανούς, που είναι η θρησκευτική ομάδα στον κόσμο που κατεξοχήν διώκεται. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Κλοντ Γιούγκερ, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω την εντύπωση ότι υπάρχει κάτι ε, που έχω να προσθέσω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω απλώς την Αυστριακή Προεδρία και σε ό,τι αφορά αυτά που υπόθηκαν για τη μετανάστευση και την πολιτική της Αυστριακής Προεδρίας. Εγώ μιλώ όχι μόνο εξ ονόματός μου, αλλά και εξ ονόματος ε, της ε, Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής συνολικά. Και όσοι πιστεύουν ότι όλα αυτά δεν ανήκουν σε μια δημοκρατική συζήτηση πλανώνται. Πάντως έχω να πω ότι υπήρξε μια ρεαλιστική προσέγγιση. Το βλέπουμε και από τα αποτελέσματα της Αυστριακής Προεδρίας. Και μπορούμε να πούμε ότι στην ε, σύντομη ιστορία των Προεδριών της Ένωσης η Αυστριακή Προεδρία θα μείνει σαν μία από τις πιο επιτυχημένες και γι' αυτό σας ευχαριστούμε. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε Ταγιάννη, αξιότιμες κυρίες και κύριοι. Δεν μου μένουν πολλά να πω. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνεργασία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα θετικά λόγια σας σήμερα. Πραγματικά υπάρχει συμφωνία που μας ενώνει σε πολλούς σημαντικούς τομείς και πολύ λίγα είναι αυτά τα οποία μας χωρίζουν. Σίγουρα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, τις ακούσαμε, αλλά και μεταξύ των ομάδων να εκπροσωπούνται διαφορετικές απόψεις. Αυτό είναι το οποίο διαμορφώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαμορφώνει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Παρά όμως τις διαφορές και τις ενδεχόμενες διαφωνίες, είναι σημαντικό να προχωρήσουμε από κοινού ε, και να προβούμε στις αλλαγές και στις μεταρρυθμίσεις, τις οποίες θεωρούμε ότι είναι σημαντικές. 28 κράτη-μέλη, τρία θεσμικά όργανα πολύπλοκα και η συνεργασία πολύπλοκη. Είμαι σίγουρη ότι καταφέραμε να σημειώσουμε πρόοδο και για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο με 53 τριμερεί διαλόγους και νομίζω ότι τουλάχιστον σε επίπεδο συμβούλου καταφέραμε να καταλήξουμε σε ομοφωνία. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην Ρουμανική Προεδρία που παίρνει τη σκητάλη. Σα ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δέσμευση αυτή που αναλάβατε την προσπάθεια. Διακόπτουμε για μερικά λεπτά τη συνεδρίαση. Πριν την πανηγυρική συνεδρίαση για την 20η επέτειο του ευρώ. Και τώρα, στην πανηγυρική μας συνεδρίαση για να γιορτάσουμε την 20η επέτειο από τη γέννηση του ενίου νομίσματος, του ευρώ. έξι και πήγα με την γιαγιά μου στο ανταλλακτήριο συναλλάγματο για να αλλάξω τα φράγκα μου σε ευρώ. Ε, το δωράκι που πήρα για το πρώτο μου δοντάκι. Και αυτό ήταν και το πρώτο μου χαρτζηλίκι. Θυμάμαι ακριβώ πόσο απογοητευμένο ήμουν όταν αντί για το πολυπόθητο πρώτο μου ρολόι πήρα ε, κέρματα, σε ευρωκέρματα ω μπουναμά. Ε, θυμάμαι όταν πήγα για ψώνια με τη μητέρα μου, προσπάθησε να χρησιμοποιήσει ένα καρότσι και δεν είχε ευρώ. Τότε χρειάστηκε να πάρει ένα ευρώ η μη αναστρέψιμη διαδικασία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για μια πιθανή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος. Πώς είναι δυνατόν να επενδύσετε, να κάνετε επενδύσεις, να, το, να αποταμιεύσετε χρήματα, να ανοίξετε επιχείρηση, αν δεν ξέρετε ποια είναι η συναλλαγματική ισοτιμία, που μπορεί να κυμαίνεται μέχρι και 10%. το ευρωπαϊκό νόμισμα θα ονομαστεί ευρώ. Εγκρίνεται το ψήφισμα. Η εισαγωγή των χαρτονομισμάτων και κερμάτων σε ευρώ σηματοδοτεί το πιο σημαντικό, το, ένα από τα σημαντικότερα, αν όχι το πιο σημαντικό βήμα στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Έχουμε 300 εκατομμύρια Ευρωπαίους που έχουν στην τσέπη τους το απτό σύμβολο ότι ανήκουν στην Ευρώπη. έχουμε κοινό πεπρωμένο. Το ευρώ δίνει στους καταναλωτές ε, επιλογές σε σταθερές τιμές και την δυνατότητα να κάνουν διεθνείς συναλλαγές με άλλες χώρες που επίσης χρησιμοποιούν το ευρώ. Εμένα κυρίως με διευκόλυνε στα ταξίδια, ιδιαίτερα όταν έκανα μια μαθητεία στην Ισπανία. Μπορούσα πολύ εύκολα να κάνω ανάληψη χρημάτων χωρίς να πληρώνω τραπεζικές προμήθειες και ιδιαίτερα αυτό είναι ευνοϊκό όταν είσαι κάτω των 25. Με το ευρώ όταν ταξιδεύω δεν πρέπει να αλλάξω συντάλλαγμα, δεν πρέπει να σκέφτομαι πόσο κάνει στο νόμισμα τη χώρα μου και τα τραπεζικά εμβάσματα είναι πιο εύκολα μεταξύ των χωρών που χρησιμοποιούν το ευρώ. Όταν μια ιδέα ανταποκρίνεται σε ανάγκε των καιρών, πάβει να ανήκει στο δημιουργό τη και γίνεται ισχυρότερη από του εμπνευστέ τη. Ζαμονέ. Κυρίοι βουλευτέ, Αγαπητοί φιλοξενούμενοι, σήμερα γιορτάζουμε την επέτεια των 20 ετών από το νόμισμά μας. Το ευρώ χρησιμοποιείται από 340 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες και είναι το δεύτερο νόμισμα σε σημασία στον κόσμο. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του Ευρωβαρομέτρου, τρεις Ευρωπαίοι στους τέσσερις κρίνουν με θετικό τρόπο το ενίο νόμισμα. Το ευρώ αύξησε τη διαφάνεια στην εσωτερική αγορά, αύξησε την ανταγωνιστικότητά τη, διευκόλυνε τι συναλλαγέ τι μετακινήσει στο εμπόριο και τον τουρισμό. Κατά τη διάρκεια τη οικονομική κρίση και χάρη στο, στην ποσοτική χαλάρωση που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ευχαριστώ για αυτή την πρωτοβουλία των πρόεδρων Ντράγκη, το νέο νόμισμα ε, ήταν μια σπίδα και έτσι απεφεύθη η κατάρρευση των πλέον αδυνάμων οικονομιών. Όμως, η κρίση έδειξε ότι δεν είχε οικοδομηθεί πλήρω το οικοδόμημα του ευρώ και ότι υπήρξαν και κάποια ασφάλματα όσον αφορά τη διαχείριση του προβλήματο του δημοσίου χρέου γνωστοποιήθηκε ότι θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι όλοι πεπισμένοι για την εύρυθμη λειτουργία του ενίου νομισματος και στην αίθουσα εδώ υπάρχουν συνάδελφοι που επικρίνουν το οικοδόμημα του ευρώ και θεωρούν τη λιτότητα σαν τροχοπέδι στην απασχόληση και την ανάπτυξη και το ενίο νόμισμα. Εγώ είμαι πεπισμένος προσωπικά ότι είναι θετικό το εγχείρημα του ευρώ. Αλλά το ευρώ δεν μπορεί να είναι ένας αυτοσκοπός. Θα πρέπει να είναι ένα εργαλείο ως μιας οικονομίας κοινωνικής της αγοράς. Με στόχο να δώσει ευημερία και εργασία σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι λοιπόν επιτακτικό να ολοκληρωθεί το οικοδόμημα που ξεκινήσαμε να κατασκευάζουμε. Η Τραπεζική Ένωση και η Κεφαλαιοκική Ένωση θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να ολοκληρωθούν. ...όπως θα πρέπει να προωθηθεί η Φορολογική Ένωση και η Οικονομική Ένωση δεν μπορούμε να παραμείνουμε εν το μέσο της οδού. Εκεί διακινδυνεύουμε να ε, ανατραπούμε από μια νέα κρίση, να συγκλονιστούμε από αυτή. Τα πλέον πρόσφατα στοιχεία δείχνουν μια μείωση του ρυθμού αναπτύξεως και της βιομηχανικής ε, παραγωγής. Ελοχεύει ο κίνδυνος μιας νέας έφεσης σε κάποιες ευρωπαϊκές ε, χώρες. Αναπτύσσονται, αυξάνονται κοινωνικές και οικονομικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων περιοχών της Ευρωζώνης και σε κάποιες περιοχές ένας νέος στους δύο δεν μπορεί να βρει δουλειά. Αυτό είναι απόλυτα απαράδεκτο. Είναι προφανές ότι λείπουν ακόμα αποτελεσματικά εργαλεία για επαναπρόθεση των επενδύσεων και για στήριξη της πραγματικής οικονομίας, να δημιουργηθούν στις απασχόλησεις και να τονωθεί η κοινωνική και η περιφερειακή σύγκληση. Συνεπώς, κατεπηγόντως πρέπει να δώσουμε συνέχεια στο αίτημα αυτού του Κοινοβουλίου για έναν επαρκή προπολογισμό που θα ανταποκρίνεται σε αυτές τις προκλήσεις. Έκκληση απευθύνω είναι ότι σήμερα να μην είναι μια, ένας απλός εορτασμός η σημερινή ε, ημέρα, αλλά θα πρέπει να δούμε και ποια προβλήματα παραμένουν εκρεμή. Θέλω να επομιστούμε τις ευθύνες μας. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, να επομιστούν τις ευθύνες τους και να γίνουν γρήγορα οι αναγκαίες αλλαγές για να ενισχυθεί το ευρώ, να επαναπροωθηθεί η απασχόληση και η ανάπτυξη και στο τέλος να δώσουμε στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό πολιτών εργασία, διότι χωρίς εργασία δεν υπάρχει ελευθερία, χωρίς εργασία δεν υπάρχει αξιοπρέπεια. Δίνω το λόγο στον κύριο Τρισέ τώρα, πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έχετε το λόγο κύριε Τρισέ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Τέο Πρόεδρε του Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Πρόεδρε τη Ευρωομάδα, αγαπητοί Πρόεδροι ε, των ομάδων των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων, ε, αγαπητέ Μάριο Ντράγκη, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος. Θυμάμαι τον Βιμ Ντάζεμπεργκ, τον προκάτοχό μου, που ήταν τότε αυτός που πρωτοστάτησε στην εισαγωγή του ευρώ και έχω στο μυαλό μου και το τι έγινε στο Κοινοβούλιο από το 2003 στο 2011. Ε, όποτε ερχόμουν στην Ολομέλεια πάντοτε, όπως και σήμερα, η καιρή ήταν συναρπαστική, γεμάτη προκλήσεις. Όπως και τώρα, επαναλαμβάνω, θέλω να τονίσω τέσσερις επιτυχίες του ευρώ. Πρώτον, επιτυχία σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την σταθερότητα του νομίσματος. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από ευρωπαϊκή δημοκρατία έλαβε την πρωταρχική εντολή της προστασίας σταθερότητας των τιμών και από την σύλληψή της ε, έκρινε το πώς μπορεί να ορίσει τις ε, τιμές και ετέθη ε, ε, και το 1,75% σε ό,τι αφορά ε, τον πληθωρισμό. Κάτι πιο θετικό σε σχέση από ότι τα εθνικά νομίσματα του παρελθόντος. Η σταθερότητα του ευρώ αντικατοπτρίζεται και στη διεθνή αξιοπιστία του νομίσματος. Είναι το δεύτερο πιο σημαντικό νόμισμα στον κόσμο μετά το δολάριο και ξεπερνά κατά πολύ το γεν που είναι στην τρίτη θέση. Δεύτερον, το ευρώ και η ευρωζώνη απέδειξαν ότι είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στους κραδασμούς ε, της οικονομικής κρίσης ε, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τη σημαντικότερη που έπληξε την Ευρώπη. Το ενιαίο νόμισμα ε, κάποιοι θεωρούσαν ότι δεν θα επιβιώσει, όμως οι εμπνευστέ του ήταν πραγματικά τολμηροί, ήταν οραματιστές και το ευρώ απέδειξε ότι προβλέψει ότι δεν θα μακροημερεύσει ήταν εσφαλμένες. Ε, αντιστάθηκε και υπό τις πιο δύσκολες ε, συνθήκες και περιστάσεις ε, σε διεθνές επίπεδο και σε ό,τι αφορά την σταθερότητα της Ευρωζώνης για να μην μακρηγορήσω, θα έλεγα ότι 15 χώρες που ήταν μέλη της Ευρωζώνης όταν ε, κατέρευσε η τράπεζα Lehman Brothers, εξακολουθούν βέβαια σήμερα να είναι μέλη και η Ελλάδα είναι μέλος επίσης και έχουμε επίσης και τέσσερα νέα κράτη-μέλη τα οποία προσχώρησαν μετά ε, την έναρξη της ε, φρικτής, της πιο φρικτής με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Έτσι νομίζω ότι αντικρούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα επιχείρηματα περί μη σταθερότητας και αντοχής τη Ευρωζώνης και του Ευρώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη λαϊκή υποστήριξη προς το Ευρώ, όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε Ταγιά, νομίζω ότι είναι αξιοσημείωτο το ότι το 75% τρεις στους τέσσερις συμπολίτε μας ε, εγκρίνουν ε, ε, το νόμισμα, το κοινό νόμισμα για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Και μόνο 20% των συμπολιτών μας είναι αντίθετοι. Πρόκειται για το πιο υψηλό ποσοστό από την δημιουργία ή από τότε που ε, έγινε λόγος ε, για ένα κοινό νόμισμα. Υπάρχουν ε, πράγματα που δεν λαμβάνονται υπόψη από σχολιάζουν τα τεκτενόμενα και είναι αυτά που εξηγούν και τη σταθερότητα της Ευρωζώνης και του ευρώ. Θα ήθελα τέλος να μιλήσω και στο τελευταίο data map το που δείχνει ότι δεν υπάρχει και τόσο μεγάλη διαφορά σε ό,τι αφορά ε, την αγοραστική δύναμη κατακεφαλή στη ΣΥΠΑ και στην ε, Ευρώπη. Περίπου η ίδια, ε, τα ίδια ποσοστά από τότε που το 1999 εισήχθη το ευρώ. Και επίσης πιστεύω πως